Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε λάβει από τους μεταρρυθμιστές συντηρητικούς ε, αιτήματα για αντικαταστάσεις και διορισμούς ε, στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ο κατάλογος με τις προτάσεις αυτές για τους διορισμούς και τις αντικαταστάσεις θα περιληφθεί στα πρακτικά της Συνόδου θα θεωρηθούν ως εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και ιδιορισμοί σε περίπτωση που δεν υποβληθούν να τηρήσει παρατηρήσεις πριν την έγκριση των πρακτικών. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα.